με ευφυή τρόπο. Όταν σου λέει πρέπει να πας αριστερά και εσύ πας δεξιά, τι ευφυέ σύστημα να είναι αυτό. Ευχαριστώ κυρία Γένσεν, λέει ο πρόεδρος. Η συζήτηση ολοκληρώνεται και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα, χώρα αύριο στις 12. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο θέμα, η έκθεση Στέρξ για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων πλοίων. Ο κύριος Στέρξ έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όταν ένα μεγάλο ε, πλοίο έρχεται από το Κντάνσκ της Πολωνίας στην Αμβέρσα του Βελγίου, παραμένει μέσα σε ευρωπαϊκά έδαφος και μπορεί να ξεφορτώσει μέσα. Αντίστροφα όμως από την Αμβέρσα για τον Γκτάνσκ πρέπει να περάσει από μία σειρά διατυπώσεων. Αυτό επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε προς όφελος των θαλασσιών μεταφόρων. Ε, θα ήθελα εντωμεταξύ να ευχαριστήσω του συναδέλφου από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά και όλου του συναδέλφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολύ καλή συμφωνία που επιτύχαμε. Οι κύριε γραμμέ αυτή τη συμφωνία είναι πάνω απ' όλα η απλούστευση, η διοικητική, η γραφειοκρατική, η ε, ηλεκτρονική διακίνηση των πληροφοριών και η πρόσβαση στον ε, ενδιαφερόμενο με το σύστημα το μονοθυριδικό. Ένα σύστημα πληροφορικής δηλαδή, το οποίο είναι συνδεδεμένο με όλα τα άλλα. Έτσι μπορούμε να έχουμε και ε, εξοικονόμηση κόστους. Το μόνο που δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε θα ήταν ε, η απαλλαγή για το φορτίο σε περίπτωση που το σκάφος που φτάνει στο λιμένα μας, στον ευρωπαϊκό λιμένα, έχει διέλθει από τρίτη χώρα. Αλλιώς υπάρχει απαλλαγή για το φορτίο. Υπάρχει απαλλαγή από την υποχρέωση να τυπώσουν δηλαδή αυτομάτως. Επίσης πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει και το ζήτημα των ε, εσωτερικών θαλασσιών, των εσωτερικών πλωτών οδών, δηλαδή των ποταμών, έτσι ώστε να διασυνδεθούν και με τις θαλάσσιες μεταφορές. Γλώσσα μία και ενιαία θα είναι η αγγλική για απλούστευση των διαδικασιών Δυστυχώς όμως το Συμβούλιο εκόφευσε στις ε, προσπάθειες της δικές μας και τις εκκλήσεις μας ε, στην έκκληση δηλαδή να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος επικοινωνίας προφορικής ή γραπτής για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό που εγώ εννοώ ότι πρέπει να υπάρχει μόνο μία γλώσσα χρηστική, η αγγλική δηλαδή. Το σύστημα επίση τη πλοήγηση. Όταν έρχεται ένα πλοίο σε ένα λιμένα μπορεί να έχει απαλλαγή ο πλοίαρχος από το, από το κόστος ή από τις διατυπώσεις του συστήματος πλοήγησης. Η επιστροπή μας υπόσχεται ότι θα προχωρήσει το δυνατό στην επεξεργασία και αυτού του στοιχείου για το χρονοδιάγραμμα τώρα, γιατί υπήρχε μια πρόθεση για σημαντική καθυστέρηση, για προθεσμίε που θα προκαλούσαν σημαντική καθυστέρηση. Εμεί θέλουμε το έχετε δυνατό να τεθεί σε εφαρμογή. Προτάθηκε αρχικά η 1η Ιουλίου του 2015 και μια και έχουμε ήδη προχωρήσει στην πρώτη ανάγνωση, έχουμε φτάσει δηλαδή στην πρώτη ανάγνωση, μπορούσαμε να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο ακόμα. Και Πρόεδρε, για να κλείσω, είναι πολύ σημαντικό ε, για τις εσωτερικές μεταφορές εμπορευμάτων να προχωρήσει το σύστημα αυτό είναι ταυτόχρονα πολύ σημαντικό και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μεταφορών μας. Έχουμε ήδη προχωρήσει σημαντικά. Το Συμβούλιο από την πλευρά του βλέπει μόνο δυσκολίες, δηλαδή το κόστος, χωρίς όμως να ε, ομολογεί ότι ένα νέο μέτρο μπορεί να προσφέρει και σημαντική εξοικονόμηση. Όφελος δηλαδή ε, για όλους μας. Εμείς Θέλουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να φτάσουμε σε μια εσωτερική αγορά, ολοκληρωμένη αγορά, αντίθετα από το Συμβούλιο, το οποίο κολλησιεργεί και προσπαθεί να καθυστερήσει αυτή την, ε, ε, αυτό το στόχο. Αισθάνομαι όλο και περισσότερη δυσφορία από τη στάση του Συμβουλίου, πρέπει να πω. Σήμερα που προσπαθούμε να έχουμε το ταχύτερο δυνατό ευρωπαϊκές λύσεις, το Συμβούλιο πατάει φρένο. Ε, ευχαριστώ όμως τους συναδέλφους για τις προσπάθειές τους και την καλή επιτυχία που είχαμε σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλλας έχει το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο εισηγητή, τον κύριο Στέρξ, για τις προσπάθειές του για την οδηγία για τις ε, διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για πλοία που καταπλέουν από πλέον απολυμμένες της Ένωσης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν είναι μόνο οι διατυπώσεις αυτές. Η οδηγία αυτή απο, απλουστεύει τις διαδικασίες και μειώνει το κόστος και για τα σκάφη και για τους καταναλωτές προσπαθώντας να διευκολύνει και να κάνει πιο ελκυστική την μικρή παράκτη ναυσιπλοΐα, Η οδηγία προσπαθεί να υιοθετήσει αυτό τον ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα, προσπαθώντας να επεκτείνει την ενιαία αγορά και στις ενδοευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές, απλουστεύοντας τις ε, διατυπώσεις. Οι θαλάσσιες μεταφορές υφίστανται πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες ακόμη και για πλοία που πηγαίνουν μεταξύ λιμένων της Ένωσης, μόνο μεταφέροντας εσωτερικά αγαθά. Οι συνέπειε είναι ότι οι ενδοκινοτικές θαλάσσιες μεταφορές αγαθών αντιμετωπίζουν το έξτρα διοικητικό κόστος. Ένα σημαντικό θέμα που τέθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ήταν η προθεσμία για να μπορέσουν οι λιμένες να δεχθούν την ηλεκτρονική μεταβίβαση των διατυπώσεων. Η συμβαστική πρόταση έλεγε 15 Ιουνίου του 2015. Δεχόμαστε ε, την προθεσμία αυτή ως προθεσμία υποβολής ενός ενιαία, μιας ενιαίας θηρίδας όπως αναφέρει το κείμενο ε, μέσα στην ευρύτερη γενική προσέγγιση. Επίσης είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε την ανάγκη ευρύτερου, σαφέστερου πλαισίου για τις εξαιρέσει των καποτάζ και στι πιστοποιήσεις των λιμένων. Επίσης θα ανακοινώσουμε τα ευρήματά μας στα άλλα ε, θεσμικά όργανα και θα προτείνουμε περαιτέρω δράση βάσει των ευρημάτων αυτών. Επίση, δεχόμαστε να σα ενημερώσουμε για μια άλλα μέτρα την επέκταση στις εσωτερικές πλωτές οδού των διευκολύνσεων της ενδοκινο, των ενδοκινοτικών θαλασσίων μεταφορών που προϊόντων που φτάνουν σε λιμένες εκτός Ένωσης για τη συλλογή στατιστικών και την προσαρμογή των τεχνικών διατάξεων στην οδηγία. Συμπεραίνω, εμείς υποστηρίζουμε τη συμβαστική πρόταση που πέτυχε ο εισηγητής κύριος Στρέξ και η Προεδρία του Συμβουλίου. Πρόκειται για ένα ισορροπημένο, σωστό κείμενο που βασίζεται στις γενικές αρχές που ε, δέχεται η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάλλας. Ο κύριος Γκράντες Πασκουάλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Κάλλας, η οδηγία ε, αναφέρεται στις τελωνιακές διατυπώσεις που αφορούν σκάφη που μπαίνουν ή που αποπλέον ή καταπλέον σε ένα λιμένα. Αυτό θα, η οδηγία αυτή διευκολύνει τη μικρή παράκτεια ε, τις μικρές παράκτηρες αράσιες μεταφορές και, και μειώνει τον αριθμό των ελέγχων και των φυσικών και ε, επιεγγράφου ελέγχων στα σκάφη και τα εμπορεύματα. Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση και η έλεγχη ε, γίνονται επανειλημμένα και πολλαπλά. Ο κύριος Στέρξ, τον οποίο συγχαίρω για τη δουλειά του, έκανε μια έξυπνη πολύ σημαντική δουλειά. Ω κοιόδη εισηγητή, αισθάνομαι ότι με αντιπροσωπεύει το τελικό κείμενο. Η διαδικασία πήρε χρόνο. Κλείναμε συμφωνίες μία προς μία. Εγκρίνει από την ε, Επιτροπή Μεταφορών μέχρι τον τριμερή διάλογο τον τέλη Ιουνίου. Η συνένεση μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου προχώρησε σταδιακά και θετικά. Περιλαμβάνονται σημαντικές ε, νέες προτάσεις που έχουν θετικά αποτελέσματα, όπως είπε ο κ. Στέρεξ. Ε, η θέση σε ισχύ, το, η ενιαία θηρίδα είναι θετικές προτάσεις που αξίζει να επενεθούν. Πιστεύω ότι πετύχαμε τους στόχους που, έθεσε, που θέσαμε στην Επιτροπή και ε, κατορθώσαμε γρήγορα να υπάρξει μια συμφωνία. Ευχαριστώ και τίποτα άλλο πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Η κυρία Ντέμπορα Σερακιάν έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Στέρξ. Έκανε έξοχη δουλειά όσον αφορά αυτή την έκθεση που θέλει να διευρύνει την ελεύθερη κυκλοφορία στο θαλάσσιο τομέα και για την ναυσιπλοεία εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Συμμερίζομαι το σκοπό τη οδηγία με τον εισηγητή και θα πρέπει όλε οι μεταφορέ των εμπορευμάτων μέσω των οι δατίνων πόρων θα πρέπει να απαλλαγούν από διοικητικό άχθος για να έχουμε ένα θαλάσσιο ε, χώρο ε, θαλάσσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς σύνορα. Δεν χρειάζεται μόνο συνεργασία ικανοποιητική μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων φορέων, αλλά χρειάζονται και συστήματα απλούστευσης που να εφαρμόζονται ταυτόχρονα. Αυτό είναι αναγκαίο για να είναι εύρυθμη η λειτουργία του εσωτερικού θαλάσσιου χώρου της Ευρώπης χωρίς σύνορα, ούτω ώστε οι μεταφορέ των εμπορευμάτων τη θαλασσία οδού να είναι ε, κάτι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιείται τον το τρόπο. Η εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών μεταξύ των κρατών μελών θα επιτρέψει σε μια αναψυπλοεία πιο ρευστή μεταξύ των διαφόρων λιμένων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και θα προωθηθεί η μεταφορά εμπορευμάτων τη που μέχρι τώρα είναι κάτω το 10% του συνόλου των μεταφορά εμπορευμάτων. Η προήγηση σύμφωνα εμποδίζεται από διοικητικέ ε, διαδικασίε. Τα ηλεκτρονικά συστήματα θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν, ούτως, ώστε θα μπορούν να ανταλλάσσονται ταχύτερα οι πληροφορίε. Πέραν αυτό, η λειτουργικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό για να έχουμε πραγματική διοικητική απλούστευση η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού τρόπου των αποτελεσμάτων, των πληροφοριών ε, χρειάζεται διαλειτουργικότητα από πλευρά τεχνική για να είναι αποτελεσματική ευτυχή. Όσον τη γλώσσα, η κοινή γλώσσα ε, σίγουρα θα διευκολύνει τη θαλάσσια ναυσιπλοεία στην Ευρώπη και η επικοινωνία θα είναι ταχύτερη, θα δημιουργείται μικρότερη σύγχυση και μικρότερε διοικητικέ καθυστερήσει. Ευχαριστώ, κυρία Σερακιάνη. Και τώρα το λόγο ο κύριος Μπεσέτ. Έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τον τίτλο της έκθεσης του κυρίου Στέρξ, που ίσως είναι κάπως ε, πλεονασματικός, προκύπτει μία σαφής εικόνα, μια πολιτική επιλογή να καταστεί δηλαδή πιο ελκυστικός, πιο ανταγωνιστικός, πιο αποτελεσματικός ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών που αποτελεί για μας το μέλλον μας και άρα ε, και για λόγους περιβαλλοντικούς ο καταλληλότερος τρόπος μεταφορών. Η έκθεση, και αυτό πιστεύουν όλες και οι εξασφαλίζει πρόοδο σημαντική, επιτυγχάνονται δηλαδή οι στόχοι μας, που είναι ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών να προχωρήσει κατά τρόπο πιο εναρμονισμένο, πιο ε, ομοιόμορφο, πιο απλουστευμένο και έτσι ανεπιφύλακτα θα υποστηρίξουμε την έκθεση κατά την ψηφοφορία και έτσι θα, θα προτιμούσαμε ταχύτερες διαδικασίες και πιο πολλές διεκδικήσεις ως πιο σαφείς μάλλον διεκδικήσεις για την εξασφάλιση μιας ενιαίας γλώσσας επικοινωνίας στον τομέα αυτών, στον χώρο των θαλασσιών μεταφορών. Πάντως, συμβαστικές λύσεις με το Συμβούλιο μας ε, φαίνονται αποδεκτές και έτσι αναπιφύλακτα θα εγκρίνουμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπέσετ και τώρα το λόγο θα λάβει για δύο λεπτά ο κύριος Βαντάλεν, παρακαλώ. Πρόεδρε, είναι έξοχη η έκθεση του κυρίου Στέρξ και η έκθεση αυτή επιτρέπει με συγκεκριμένο τρόπο να ωφεληθούν οι θαλάσσιες μεταφορές, να απλουστευθούν τα πράγματα. Η Επιτροπή Μεταφορών ταυτόχρονα έθεσε προτεραιότητες στις συζητήσεις όσον αφορά την ποτάμια ναυσιπλοεία. Συμφωνούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάξει έκθεση όσον αφορά την απλουστευμένη διαδικασία για τον τομέα αυτών επίση. Και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει στα συμπεράσματά της και να κάνει ομοθετικέ προτάσεις. Όσον αφορά την απαλλαγή από τις υπηρεσίες ε, τις θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ούτω ώστε να είναι πιο θεμητό ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών πλοήγησης και να είναι ποιοτικέ οι υπηρεσίες που παρέχονται. Το είπε ο κύριος Στέρξ, η Επιτροπή Μεταφορών ήθελε να χρησιμοποιηθεί μία γλώσσα και τα κράτη-μέλη επέλεξαν μία λύση σύμφωνα με την οποία η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται με πιο κοινοτικό τρόπο. Είναι ένα πρώτο στάδιο κύριε Πρόεδρε, πολύ μετριοπαθές βήμα όμως όσο θα υπάρχουν νεκροί και τραυματίες διότι είναι θύματα ενός ατυχήματος πλοίων και, δεν μπορούν να συνεννοηθούν διότι μιλάνε δύο-τρεις διαφορετικές γλώσσες φαίνεται ότι είναι αναγκαία μια κοινή γλώσσα και παραμένει και θα πρέπει να παραμείνει η αγγλική γλώσσα όσον αφορά τις θαλάσσιες και τις ποτάμιες μεταφορές. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλεν και τώρα το λόγο για ένα μισή λεπτό έχει ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέρξ για το έργο του, συγχαίροντάς τον και για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Το κείμενο που θα υποβληθεί για ψηφοφορία στην Ολομέλεια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ε, εναρμόνιση των θαλάσσιων μεταφορών και την ανταγωνιστικότητα στι θαλάσσιε μεταφορέ, δηλαδή προ τη θέμενη αξία ευρωπαϊκή, που είναι απαραίτητη εν ώψη και τη κρίση, και ταυτόχρονα προάγει ένα μέσο μεταφορών, ένα τρόπο μεταφορών πιο οικολογικό. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι όχι μόνο απαλλάσσονται τα πλοία από τι διοικητικέ διατυπώσει, γραφειοκρατικέ διατυπώσει αγωγής και ε, εισόδου και εξόδου από το λιμένα, αλλά ταυτόχρονα και ε, διασφαλίσεται καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των πλοίων. Όσον αφορά τη χρήση μιας και νέας γλώσσας που αναφέρθηκε νωρίτερα, πιστεύω ότι η συμβαστική λύση δίνει επαρκή ε, εγγύηση, δηλαδή στο άρθρο 7 αναφέρεται χωρίς να επιβάλλεται μια ενιαία γλώσσα η δυνατότητα μιας κοινή γλώσσας, χρήσης μιας κοινή γλώσσας. Ενιαία γλώσσα είναι μάλλον και κοινή ταυτόχρονα, αν και πάντως δεν προσδορίζονται συγκεκριμένε λεπτομέρειες, πράγμα που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη, διότι ε, το να μην είναι κατανοητή η γλώσσα του ενός από τον άλλον μπορεί να έχει πολύ αρνητικές και καταστροφικές συνέπειες. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκριθεί το κείμενο του κύριου Στόρεξ με τη συμβαστική. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Ξεκινούμε με τη διαδικασία των μονόλεπτων παρεμβάσεων. Η κυρία Τικάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Η οδηγία για τις διατυπώσεις ε, των σκαφών που επιβάλλονται σε σκάφη που καταπλέουν και αποπλέουν από, από κοινωτικού λιμένε διευκολύνουν τι τελωνιακέ διαδικασίε και διευκολύνουν την ηλεκτρονική ανταλλαγή με την εισαγωγή ηλεκτρονικών ε, θαλάσσιων συστημάτων καθώ και την ενιαία θηρίδα για την ενημέρωση για τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Αυτό απαιτεί συνεργασία μεταξύ των διάφορων αρμόδιων αρχών. Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο το αργότερο στις 31 12 του 2011 για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή των ε, απλοποιήσεων που εισάγει ο οδηγία αυτή στι ε, μεταφορέ εσωτερικών πλατών, πλωτών οδών για να μπορέσει η Επιτροπή να μα ενημερώσει μέχρι ποιο επίπεδο η, το River Information System είναι συμβατό με το SafeCNet, πλατφόρμα στη δεδομένων που εφαρμόζει, που χρησιμοποιεί ο οδηγία εξασφαλίζοντα και ταχύτερη ενημέρωση με την τροπολογία 9 για την χρήση του κανόνα 40 του της συμβάσεως Σόλας που επιτρέπει την χρήση των αγγλικών σαν γλώσσα κοινωνία. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Η κυρία Μέσνερ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Ο Επίτροπο μίλησε για έναν ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα. Αυτό είναι ο στόχος τον οποίο όλοι επιδιώκουμε πιστεύω και γι' αυτό είναι πολύ καλή ε, η έκθεση εξυπηρετεί το στόχο αυτών, λοιπόν. Μεγάλο ποσοστό των, επιβατικών, ε, των επιβατικών μεταφορών αλλά και των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη περνούν από τους λιμένες μας και γι' αυτό είναι απαραίτητη η εναρμόνιση και η απλούστευση των μεταφορών αυτών. Τους δύο αυτούς στόχους επιτυγχάνει η έκθεση και γι' αυτό έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο του κυρίου Στέρξ. Δυστυχώ όμω ο κύριο Στέρξ δεν μπόρεσε να επιτύχει δύο από του ε, σημαντικού για τον ίδιο στόχου που και εμά μα βρίσκουν σύμφωνου, την ε, δυνατότητα καταρχάς για την απλούστευση στην περίπτωση της πλοήγευσης, επαλλαγής πλοήγευσης και την χρήση μιας και γλώσσα που πρέπει να είναι η αγγλική ασφαλώς. Ε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε να υπάρχουν ναυάγια, να υπάρχουν ναυτικά ατυχήματα, θαλάσσια ατυχήματα, μόνο και μόνο γιατί οι ναυτικοί μιλούν διαφορετική γλώσσα. Πρέπει να έχουμε καλύτερη και πιο ε, αποτελεσματική ναυσιπλοεία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο, πρώτα και μετά στον εισηγητή. Κύριε Κάλλας. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ πολύ για τι παρατηρήσει σα, την ομόφωνη υποστηρίξη που εκφράζεται στην πρόταση αυτή. Ε, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που προχωρήσαμε με το σημαντικό αυτό βήμα τη πρόταση του κυρίου Στέρξ και πιστεύω ότι μα περιμένουν και ακόμη μεγαλύτερα άλματα στο στόχο, στον δρόμο αυτό της ανάπτυξη ενός ενιαίου χώρου των θαλασσίων μεταφορών στην Ευρώπη και χωρίς τελωνιακούς ε, φραγμούς και πιστεύω ότι θα δούμε σημαντικές προόδους ε, περισσότερο ακόμα. Τώρα μιλούμε μόνο για διατυπώσεις. Ένα σημαντικό βέβαια ζήτημα, αλλά απλώς διοικητικό ζήτημα. Όταν όμως έρθει η ώρα να απαλλαγούμε και από τις θελωνιακές διατυπώσεις, διατυπώσεις θελωνίου, που είναι πολύ πιο περίπλοκη βέβαια υπόθεση και αμφιλεγόμενη. Θα χρειαστώ πάλι την υποστήριξη σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ντίκ Στέρξ, ο εισηγητής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που συνέβαλαν στη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους και τον κύριο Επίτροπο ο οποίος επίτροπο σωστά έθεσε το δάχτυλο επί ανοιχτής ε, πληγής όσον αφορά τις τελωνιακές διατυπώσεις. Ε, το σύστημα το τελωνιακό δεν θα είναι εντελώς ξεχωριστό από το σύστημα των μεταφορών. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο επικοινωνία. Ε, για εσά, κύριε Επίτροπε, στην οδηγία προβλέπονται διάφορα, διάφορα καθήκοντα, όπω είναι η πλοήγηση. Αλλά πέραν αυτού ε, υπάρχει και ένας ρόλος που διαδραματίζουν οι λιμένες σαν κέντρα, σαν σταυροδρόμια μεταξύ θάλασσας και ενδοχώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφορε προτάσει που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι λιμενικέ εγκαταστάσει, διότι χωρί ποιοτικά λιμάνια, μια θαλάσσια μεταφ... Ε, πολιτική θρασία μεταφορών ποιοτική δεν έχει νόημα. Η πλοήγηση στα ποτάμια θα πρέπει να δημιουργήσει και άλλες σχέσεις μεταφορικές με άλλους τρόπους μεταφορών. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε και λυπάμαι μετά που δεν μπορέσαμε να πούμε ότι τα αγγλικά θα είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιείτε. Καταλαβαίνω πολύ καλά την ευαισθησία που έχει αυτό το θέμα. Κατάγομαι από μια χώρα που διεξάγεται συζήτηση όσον αφορά τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται και η χρήση της γλώσσας ε, είναι κάτι που κοστίζει μέρες συζητήσεων Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό τον πύργο τη Βαβέλ, θα μπορούσαμε να αρκεστούμε σε μία και μοναδική γλώσσα. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα συναισθηματικό, είναι ένα θέμα τεχνικό. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των δύο. Και ελπίζω, κύριε Επίτροπε, ότι θα μπορέσετε να σημειώσετε πρόοδο επί τη βάση των διαφόρων ε, προβλέψεων που περιέχει η οδηγία. Θα πρέπει να υπάρξει και επαφή με του διεθνεί ναυτιλιακού οργανισμού. Εκεί έχουν συναυθεί πολλέ συμφωνίε που είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τι ελάχιστε μεταφορέ. Και πίσω από τη γλώσσα είναι και το θέμα το ανθρώπινο. Η χρήση της γλώσσας είναι κάτι σημαντικό. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη του θαλασσίου τομέα που θα είναι σίγουρος, αποτελεσματικός, ασφαλής και που θα σέβεται και το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλό κουράγιο και ε, θα πρέπει παρακαλώ να λάβετε υπόψη αυτά που ζητούμε μέσα στα πλαίσια του άρθρου 11α αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, έληξε συζήτηση. Θα γίνει ψηφοφορία αύριο στις 12. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Gross